No, can you write, can you write it down here? Thank you, with big... Hello everybody. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στην συνεδρία της Επιτροπής για σήμερα. Anybody wants to take the floor already? Κάποιο ζητάει ήδη το λόγο, λέει προεδρό. Θέλετε να με αντικαταστήσετε, όχι πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Χθε λάβαμε τον κατάλογο τη ε, ψηφοφορία στι 6 το απόγευμα. Βρισκόμαστε σε μια επιτροπή που ασχολείται με θέματα απασχόλησης. Γι' αυτό λοιπόν το θεωρώ απαράδεκτο να λαμβάνουμε κατάλογο ψηφοφορία στις 6 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν βοηθοί οι οποίοι εργάζονται βράδια. Ε, θέλουμε, λέμε, να έχουμε ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, καλά ωράρια, αλλά θεωρώ απαράδεκτο το να λαμβάνουμε 6 ώρα το απόγευμα κατάλογο ψηφοφορίας, ε, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη μέρα το πρωί, για τον οποίο έχουν δουλέψει βράδυ άτομα. Αυτά, ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ μαζί σας, λέει η Πρόεδρος. εγώ άνοιξα τον ε, κατάλογο και δεν ήξερα καν ούτε εγώ τι είχαμε μπροστά μας. Είναι πάρα πολύ αργά να το λαμβάνουμε στις 6 ε, ώρα το απόγευμα, ε, ιδιαίτερα για τις ομάδες. Θα βοηθούσε όλους μας, λέει Πρόεδρος, και ιδιαίτερα τους βοηθούς των πολιτικών ομάδων, να λαμβάνουμε τους καταλόγους νωρίτερα. Λοιπόν, όλες οι γλώσσες της Επιτροπής μας είναι διαθέσιμες σήμερα εκτός των Μαλτέζικων, λυπάμαι, συνάδελφε, αλλά είστε μοναδικός, είστε μοναδικός. Έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για το Κοινωνικό Ταμείο Plus και χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία προκειμένου να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Πέραση ψηφοφορίας. Adopted. Ενεκρίθη. Yes. Any problems, technical problems? Έχουμε ε, κύριε Αντατσόφσκι, υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Ωραία, συνεχίζουμε. Σημείο 5, πρώτος κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού 1309, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψήφος υπέρ. Ζητώ συγγνώμη. Η ηλεκτρονική είναι η ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία ή η ηλεκτρονική λέει τώρα η πρόεδρος. Have you all voted? The vote is closed. Πέρας. Είναι κρίθη. Item 6. Σημείο 6 πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικές της Ευρωζώνης. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε ηλεκτρονική ψήφο, έχουμε τη συμβαστική 5, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές. Συμβαστική 6, ναι, εγκρίνεται. Συμβαστική 6, Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Ονομαστική ψήφο ζητάει το ΕΛΚ. Το SND με συγχωρείτε. Για το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. 86. 86, δεύτερο τμήμα. Vote open. Have you all voted? Πέρα στις ψηφοφορίες. εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2β τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ. Everybody voted. Vote is closed. Peras. Carried. Amendment 100. Who is... Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά αποχές ασαφές, λέει ο Πρόεδρος. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Everybody votes it. Vote is close. Πέρας. 26 to 21 carried. 26 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται. Καλώς λέει τώρα η Πρόεδρος εναντί σχολείου που δεν έχουμε ακούσει. Άρχεται η ψηφοφορία. Everybody voted. Vote is closed. ψηφοφορίας. Carried. Εγκρίνεται. 108. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Παρακαλώ, ψηφίστε. Have you all voted? Vote is closed. Ψηφίσατε, πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ Vote is open. Everybody voted. Vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται 147 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Everybody votes it. Vote is close. Πέρας, παρακαλώ. Εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 172 πέραν της συμβαστικής 22 ως συμπληρωματική δηλαδή υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα 181. Δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε, παρακαλώ. Everybody Απορρίπτεται. 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 186. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189. Υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε εδώ την 189 παρακαλώ πέρας απορρίπτεται συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 λέει η πρόεδρος, συμβαστική 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 208 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία η 208 μάλιστα ψηφίσατε πέρασε απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 209 παρακαλώ πέρας απορρίπτεται συμβιβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.11 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ ψηφίστε πέρας εγκρίνεται 2.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αναφορές 1 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ πέρας εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έξι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επτά, υπέρ, κατά α, αποχής εγκρίνεται. Επτά. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οκτώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δέκα. Υπέρ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 αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Everybody voted, vote is closed. Εγκρίθηκε 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ. Καλά, κατά, με συγχωρείτε, <laughs> αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ προφορική του S&D υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μου ζητάνε να ελέγξω. Οκ, ψηφίζουμε. Για την 31. Rejected. Απορρίπτεται. Άρα δεν έχουμε την προφορική πλέον. Ναι, δεν έχουμε την προφορική, λέει η Πρόεδρος. Amendment 32. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Προφορική. Του S&D. Προφορική του S&D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Τη 43 παρακαλώ ψηφίστε. Have you all voted or is... Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. «48» είπε η Πρόεδρος, ο Διερμηνέας είπε σωστά το 49, τώρα το 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμμεθική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 59 παρακαλώ ψηφίστε δεν Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 που είναι προφορική του S&D. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Την 68 παρακαλώ. Voted. Πέρασε. 69 in favor. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορι... Ε, εγκρίνεται, με συγχωρείτε. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική τελική ψήφος. Παρακαλώ. Have you all voted? Vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. or what? Uh, uh, so let me, let me congratulate. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την κυρία Τόμ, η συγγήτρια. Get to the European Court of Auditors Special... Περνάμε στην ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για το Ταμείο Βοήθειας στους Απόρους. Θα παρακολουθήσουμε μία παρουσίαση για ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα. Η παρουσίαση θα είναι γεμάτη στοιχεία και μια που μ' αρέσει να βλέπω στατιστικά στοιχεία θα σας παροτρύνω να μείνετε για να παρακολουθήσετε την παρουσίαση και είμαι σίγουρη ότι θα σας χρησιμεύσουν πάρα πολύ όσα θα ακούσετε. Whoever is not interested in the presentation... Όποιος δεν ενδιαφέρεται για την παρουσίαση, παρακαλώ να αποχωρήσει από την αίθουσα. So let me welcome uh, our guests from the να καλωσορίσω λοιπόν τους προσκεκλημένους από το Ελεκτικό Συνέδριο. Καλώς ήρθατε. Δεν γνωρίζετε, όμως εκτιμώ πολύ τις εκθέσεις σας, διότι πάντα είναι γεμάτες πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για θέματα τα οποία συζητάμε πολύ εδώ στην Επιτροπή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα στοιχεία, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξεις κάτι και να οδηγηθείς σε σωστά αποτελέσματα. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για 10 λεπτά για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας και ε, να κάνετε μία σύντομη παρουσίαση. Κατόπιν θα δώσω το λόγο του στους συντονιστές και στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για τυχόν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι ενώπιον της Επιτροπής Απασχόλησης ε, και μένα μου αρέσει πολύ η Επιτροπή σας ε, και εκτιμώ το έργο σας διότι ήμουν εισηγήτρια στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία αρκετών εκθέσεων ε, για παράδειγμα της έκθεσης για την απασχόληση των νέων. Είχαμε παρουσιάσει τρεις εκθέσεις του συνεδρίου ε, για ε, το θέμα αυτό και για την ενσωμάτωση των ε, μεταναστών, για άλλα θέματα, για την παιδική φτώχεια, την μακροχρόνια ανεργία. Όμως σήμερα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε την έκθεση σχετικά με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να εκπροσωπήσω το τμήμα 2 του ελεκτικού συνεδρίου ως αντικαταστάτρια του εισηγητή, ο οποίος ε, έχει αποχωρήσει από το ελεκτικό συνέδριο. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά ε, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια στην αρχή. Παρά τον πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ακόμα ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους που κινδυνεύει ε, με κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της φτώχειας. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ο στόχος είναι ε, να βγουν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2020 ο κίνδυνο είναι μεγαλύτερος για συγκεκριμένε ομάδες όπως παιδιά και ηλικιωμένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει διαθέσει 3,8 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους ε, για την περίοδο 2014-2020. Ο στόχος του Ταμείου είναι η απα... είναι η διόρθωση, είναι να... Ε, η προσπάθεια να βγουν από τη φτώχεια αυτά τα 20 εκατομμύρια Ευρωπαίων. Σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, το Ταμείο αυτό έχει ε, επιφέρει ορισμένε αλλαγές. Καταρχάς, προσφέρει και ηλική βοήθεια και ε, μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο ξεχωριστών προγραμμάτων το τύπου 1 και τύπου 2 και θα υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης κονδυλίων από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να συνεχίσουν με περισσότερες ε, λεπτομέρειες και επεξήγηση των διαφανειών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ιβάνοβα, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήμουν υπεύθυνο του ελέγχου και της ομάδας που τον ε, διεξήγε. Πρόκυψαν τα εξή ερωτήματα, λοιπόν. Καταρχά, ε, θέλαμε να μάθουμε αν το νέο ταμείο ήταν, είναι αποτελεσματικό για την καταπολέμηση τη φτώχεια. Χωρίσαμε λοιπόν σε τρεις κύριους θεματικούς άξονες την ε, έρευνά μας. Ε, πρώτον, το ΦΕΑΝΤ αντικαταστάτη του προηγούμενου προγράμματος. Το αν το ε, ταμείο μπορεί να βοηθήσει με στοχευμένη βοήθεια και εάν τα μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης μπορούν να επιφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον έλεγχο. Όταν γίνεται λόγος λοιπόν για το ταμείο αυτό, το ΦΕΑΝΤ, να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά ε, δύο ξεχωριστέ κατηγορίε προγραμμάτων. Το, η κατηγορία 1 και η κατηγορία 2, OP1. Ε, επιχειρησιακά προγράμματα 1 επιχειρησιακα προγραμματα 1 λοιπον και επιχειρησιακά προγράμματα 2. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 1 παρέχει κυρίως επιστημιστική βοήθεια. Βλέπουμε εδώ ότι το 90% της επιστημιστικής ε, βοήθειας διανέμεται σε πέντε κράτη-μέλη. Την Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ισπανία και 2,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου πηγαίνει στα επιχειρησιακά προγράμματα τύπου 2, τα οποία παρέχουν μια πιο ε, στοχευμένη προσέγγιση για την ε, κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. Τα ευρήματά μας λοιπόν έχουν ως εξής. Συνδυάσαμε διάφορες ενδυμασίες έρευνες και είδαμε ότι το Ταμείο είναι γενικά ευπρόσδεκτο από τους δικαιούχους. Όμως ε, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για το πόσο σημαντικό είναι. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα στα κράτη-μέλη και λίγες σχετικά ενδείξεις για τη σημασία του Ταμείου. Το Ταμείο αυτό παρέχει περισσότερες ε, δυνατότητες από το προηγούμενο, διότι έχει νέα μέτρα και δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση όταν εφαρμόζουν μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αυτό λοιπόν είναι μια καινοτομία του ΦΕΑΝΤ. Η έρευνα εστάλει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έτσι ώστε να αποκομίσουμε μία εντύπωση της ε, σημασίας τους. Δυστυχώς ελάχιστα κρατημέλη μας απάντησαν, όπως όμως από τις απαντήσεις είδαμε ότι είναι αρκετά ορατό σε θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης ε, και βοήθειας προς τους απόρους. Η ορατότητά του είναι περίπου 5-10% στο Λουξεμβούργο και υπάρχουν χώρες όπως η Πολωνία όπου ε, η επιτυχία αγγίζει το 67%. Αυτά είναι βέβαια μόνο ενδείξεις της ε, συνολικής δύναμης του Ταμείου αυτού. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μία εκτίμηση της γενικότερης εικόνας του ΦΕΔ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα τύπου 1 επισητιστική βοήθεια δηλαδή, υλική βοήθεια και τα συνοδευτικά προς αυτά μέτρα προς τους απόρους. Εξετάσαμε συνολικά εννέα προγράμματα και είδαμε ότι οι ομάδες τις οποίες στοχεύουν διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Ε, μάλιστα βρήκαμε αρκετά ευρύς ορισμούς για το τι καθιστά ε, άπορο, έναν άπορο το κάθε κράτος μέλος λοιπόν έχει διαφορετική αντίληψη. Συνειδητοποίησαμε ότι τα μισά κρατημέλη συνδέουν το ταμείο αυτό με κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας ε, τα οποία έχουν σχέση με, τις, ε, με την κοινωνική πρόνοια. Ο ορισμός βέβαια του ε, απόρου όπως σας είπα, διαφέρει. Από τη μία βλέπουμε ότι κάποιοι άλλοι φορείς ε, είναι αρμόδιοι για να καθορίσουν ε, τις ε, παραμέτρους, σε κάποια, ε, σε κάποια άλλα κράτη-μέλη γίνεται κεντρικά, με κρατικές δομές. Αναφέρθηκα τώρα σε συνοδευτικά μέτρα. Τα συνοδευτικά μέτρα είναι υποχρεωτικό κομμάτι των, της βοήθειας που παρέχουν τα κράτη-μέλη υπό το ΦΕΑΝΤ. Αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να παρέχουν βοήθεια με τη μορφή ενημέρωσης φυλαδίων, έτσι ώστε να ενημερώνονται οι δικαιούχοι για τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εκείνους, ιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές κτλ. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα υποχρεωτικά μέτρα, όμως είναι δύσκολο να γίνει μια σύγκριση διότι ε, διαφέρουν ως προς ε, τον ε, τρόπο προβολής. Γι' αυτό και δεν έχουμε κοινού δείκτες για την απήχηση των συνοδευτικών αυτών μέτρων. Σε γενικές γραμμές είδαμε ότι ότι ο έλεγχος της ε, σύνδεσης των ε, προγραμμάτων με το ΦΕΑΤ μπορεί να γίνει υπό τα προγράμματα της κατηγορίας 1, δηλαδή της επιστικής βοήθειας, αλλά και ε, της κατηγορίας 2, η οποία αποτελείται κυρίως από προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Χρειάζεται όμως ε, να καταβληθεί με μεγαλύτερη προσπάθεια έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις συνδέσεις ε, του Ταμείου αυτού με το ESF. Τώρα, πού στοχεύουμε. Καταρχάς, να βελτιώσουμε την διαδικασία επιλογής ε, δικαιούχων. Ποιος δηλαδή δικαιούται να λάβει βοήθεια από αυτό το ταμείο, ποιες είναι οι ομάδες και υπό ποιες προϋποθέσεις. Έπειτα, θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικό να υπάρχει καλή συνεργασία με τους συνεργαζόμενους φορείς. Γι' αυτό χρειάζεται ένα κοινό πλαίσιο το οποίο θα καθοδηγεί τους φορείς αυτούς. Έπειτα, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγουν μια ε, ολοκληρωμένη αξιολόγηση του ε, ΦΕΑΔ για να βγουν πορίσματα σχετικά με το πώς μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική ενσωμάτωση. Γι' αυτό φυσικά χρειάζεται και η συνεργασία των ε, διαφόρων φορέων από τους οποίους εξαρτάται εν μέρει η επιτυχία του Ταμείου. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ξεκινάμε από τους συντονιστές. Ε, δεν ξέρω αν ε, εσείς ή κάποιος αντικαταστάτης σας θέλει να κάνει ερώτηση. Από το ΕΛΚ πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρατήρησα ότι αναφερθήκατε κυρίως στην επισητιστική βοήθεια ως ε, κύριο ε, στόχο του προγράμματος. Η συνεισφορά του Ταμείου στην μείωση της φτώχειας δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα με μετρήσιμα μεγέθη. Χρησιμοποιείται μεν το Ταμείο για επισητιστική βοήθεια, όμως ε, αυξάνονται οι ανάγκες και αυξάνεται και το ποσό χρηματοδότησης. Εμείς βέβαια πρέπει να κάνουμε προσπάθειες ε, για να μειώσουμε την ε, φτώχεια. Ας μην ξεχνάμε όμως τη σημασία που έχει η επιστημιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντηση προς την ε, έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου αναφέρει ότι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της ε, φτώχειας είναι η καταπολέμηση των ε, αιτίων και γι' αυτό χρειάζεται επισητιστική βοήθεια μαζί με συνοδευτικά μέτρα και κατάλληλη καθοδήγηση των ε, ευάλωτων αυτών ομάδων, των παιδιών κτλ. για τις δυνατότητες που έχουν, για υπηρεσίες υγείας κτλ μέσω του EMFF και του ESF Plus μπορούμε να εστιάσουμε στις πιο ευάλωτες ομάδες της ε, κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ESF ε, Plus θα πρέπει να επιμείνουμε να αυξηθεί ο προσυπολογισμός του ESF Plus κατά 3% έτσι ώστε να περιλαμβάνει και ειδικά μέτρα για κοινωνική ενσωμάτωση. Νομίζω πως ε, είναι κάτι που μπορούμε να στηρίξουμε, διότι δεν πρέπει να, φύ, να παρατήσουμε στο έλεος του Θεού τους ε, πιο ευάλωτους αυτής της κοινωνίας. Μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, αλλά θα ήθελα να πω ότι Είδατε λίγο τα αρνητικά ίσως της έκθεσης. Μπορείτε ίσως να το συνδυάσετε και με άλλες εκθέσεις που έχουμε και τότε θα έχετε μια άποψη πιο θετική. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι σε αυτή την έκθεση περιλαμβάνονται καλά νέα παρά τις επικρίσεις. Παρά το ότι πάνω από το 83% της χρηματοδότησης του Φέα διατίθεται ακόμα για επισητιστική βοήθεια. Αυτό είναι γεγονός, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, αλλά έχει γίνει μεγάλη πρόοδος προς ε, μέτρα κοινωνικής ένταξης. Αυτό που μένει είναι να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά στο μέλλον. Στην, ε, ε, δεν θέλαμε να μετρήσουμε την εφαρμογή, αλλά περισσότερο να δούμε τι έχει γίνει με τον σχεδιασμό σε σχέση και με το προηγούμενο πρόγραμμα που υπήρχε πριν. Έχετε δίκιο ότι οι πιο ευάλωτε ομάδε θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αλλά γι' αυτό κάναμε και τι συστάσει, για να υπάρξει καλύτερη στόχευση. Γιατί μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε πώς έχουν επηρεαστεί αυτές οι ευάλωτες ομάδες. Ναι, διαθέσαμε χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες. Αλλά δεν έγινε αυτό απαραίτητα με τον πιο αποδοτικό οικονομικά τρόπο. Γιατί, Γιατί δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε αποδείξεις. Και γι' αυτό κάναμε την πρώτη μας σύσταση, καλύτερη στόχευση, να ορίσουμε καλύτερα ποιες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες. Όχι γιατί σπαταλήσαμε χρήματα, αλλά γιατί αυτά τα χρήματα ίσως δεν διατέθηκαν για τις ανάγκες που τα είχαν περισσότερη ανάγκη. Ο κύριος Πάτεν, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την έκθεση. Είμαι καινούριο εδώ στο Κοινοβούλιο και είπε η πρόεδρος αν ενδιαφέρεται για τα δεδομένα. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομεί εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο που έχουν ανάγκη από αυτά τα στοιχεία. Βρίσκω λοιπόν άριστη την έκθεσή σα. Θα ήθελα όμω να κάνω και κάποια σχόλια. Πρώτον, καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι υπάρχουν καλά νέα σε αυτή την έκθεση, αλλά υπάρχει κάτι όσον αφορά την συμβολή για την μείωση της φτώχειας που δεν έχει αποδειχτεί και ότι υπάρχουν ε, ακόμα 4,5 εκατομμύρια λίρες σε αυτό το πρόγραμμα που μένουν να δαπανηθούν. Όταν λέτε ότι το 83% λοιπόν της χρηματοδότησης διατίθεται για τρόφιμα και το 90% διατίθεται σε πεντε κράτη-μέλη, εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τις συστάσεις σας, Είπατε ότι χρειάζεται παρέμβαση, αποτελέσματα, μίλησατε για στόχευση και μεθοδολογία. Έχω να κάνω μια υπόδειξη. Έχω δουλέψει σε αυτόν τον τομέα και συμμετείχα στην εφαρμογή ε, κονδυλίων, ταμείων κτλ. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου ως μέρος του προγράμματος και αυτό να προβλεφθεί ήδη από την αρχή. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τα κράτη-μέλη και τους εταίρους τους να μας πούν εκ των υστέρων πώς είχαν τα πράγματα. Θα πρέπει ήδη από πριν να έχουμε μια ευρεία μεθοδολογία, όλοι να συμβάλλουν και να ε, μπορέσουμε έτσι να εκτιμήσουμε ε, τον αντίκτυπο. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Εγώ βρήκα μία από τις προηγούμενες εκθέσεις ε, της Επιτροπής ένα έγγραφο εργασιών αξιολόγησης ε, ήταν πραγματικά εκπληκτική δουλειά. Όλα ήταν ξεκάθαρα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε από την προπαγάνδα και να, γίνουμε, ε, να υιοθετήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα είναι πολύ περισσότερο προσβάσιμο εάν οι μικρότερες οργανώσεις, οι εταίροι των ε, κρατών μελών μπορούν να έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να πλουστευτεί η διαδικασία. Και κυρίως, το ταμείο αυτό έχει να κάνει με την αηφορία. Θα ήταν λοιπόν πολύ καλό ναι, σε επίπεδο κράτους μέλους να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια με τη διανομή τροφίμων, αλλά θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τους τοπικούς οργανισμούς που διανέμουν τα τρόφιμα, ούτω ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Νομίζω ότι θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στην τοπική αηφορία. Και, όπως είπε και η Πρόεδρος, αυτό που μας απασχολεί είναι τι θα γίνει μετά, γιατί θα ενσωματωθεί το Ταμείο στο ESF+. Και έχω κάποια ερωτήματα όσον αφορά αυτό. Απρόβλεπτες συνέπειες, για παράδειγμα. Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, ναι, έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Διότι οι τοπικοί οργανισμοί κάνουν κάτι καλά, δεν τα κάνουν όλα καλά. Όσον αφορά λοιπόν την ενσωμάτωση με το ESF, είναι καλό να θέλουμε να τα συγχωνεύσουμε όλα. Αυτό το πρόγραμμα έχει να κάνει με την κοινωνική ένταξη και τον επισητισμό. Ίσως λοιπόν να πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, δηλαδή τρόφιμα και υλική βοήθεια και όσον αφορά την κοινωνική ένταξη αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Πρόεδρος, Λυπάμαι πολύ, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε ότι κάθε ερώτηση θα πρέπει να διαρκεί μόνο δύο λεπτά. Γίνεται μια συζήτηση αυτή τη στιγμή και τώρα το λέω ξεκάθαρα, θα είναι καλό για όλους και για τους καλεσμένους μας, μόνο δύο λεπτά χρόνος ομιλίας από εδώ και μπρος. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, μάλλον ποιος θα απαντήσει στον κύριο Πάτεν, η κυρία Βάνοβα. Είπα ότι και άλλοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Θέλετε πρώτα να μιλήσουν όλοι και μετά να απαντήσουμε. Ναι, συμφωνείτε σε αυτό, ρωτάει η πρόεδρο. Συμφωνούμε λοιπόν, με τις, ε, προχωράμε με τις ερωτήσεις. Ο κύριος Μίλλερ, στη συνέχεια, Γκουίντο Ράιλ, όχι τώρα, απλώς διαβάζω τη λίστα των ομιλητών. Κυρία Ραφάλσκα, κύριος Μπίλκουες, Σαλάνη, Μαρίνο και ο κύριος Μίλλερ τελευταίος και η κυρία Λάγκεν Ζίπεν στη συνέχεια. Κύριε Ράιλ. Ευχαριστώ πολύ. Είδα και εγώ την έκθεση και με μεγάλη μου χαρά είδα ότι ασχολείστε και με το θέμα των αστέγων. Με σοκάρει πόσους άστεγους βλέπουμε στους δρόμους ευρωπαϊκών πόλεων και κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Είμαι τρεις μήνες ευρωβουλευτής και Κοιτάζω έτσι γύρω στις Βρυξέλλες και μου κάνει τρομερή εντύπωση το τι συμβαίνει. Ε, βλέπω όμως και στη Γερμανία, στο Μόναχο, στο Βερολίνο, το, Αμβούργο, το Αμβούργο, στη γειτονιά μου, στη δική μου πατρίδα, στην περιοχή του Ρούρ. Βλέπω ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, υπαρκτό και πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι οι οποίοι έχουν ε, διάφορες, ε, πάσχουν από ψυχικές ασθένειες. Υπάρχουν άστεγοι από χώρες της ε, πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Ε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ε, βρίσκεται κάποιος στο δρόμο. Στη Γερμανία μπορεί να βρεθεί κάποιος στο δρόμο απλά επειδή ε, τα νίκια είναι υπερβολικά ακριβά και δεν κερδίζει αρκετά με την εργασία του. Προσπαθήσαμε στη Γερμανία να ελέγξουμε κάπως την κατάσταση, αλλά το πράγμα είναι πραγματικά ανεξέλεκτο. Έχουμε υποτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος, ε, νομίζω. Υπάρχουν ε, διάφορες προγνώσεις που μόνο αρνητικές τάσεις δείχνουν. Γι' αυτό λοιπόν Έχω εγώ μία συγκεκριμένη ερώτηση. Στη Γερμανία το πρόβλημα είναι τεράστιο, γιατί λοιπόν η Γερμανία λαμβάνει ένα κλάσμα ένα μελιτέο ποσό από το σύνολο του διαθέσιμου ποσού του Ταμείου, δεδομένων των ε, προβλέψεων και των στοιχείων που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ραφάλσκα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Είναι καλό το ότι υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες εδώ, δηλαδή Υπάρχουν, ε, υπάρχει διανομή τροφίμων και επίσης η κοινωνική ένταξη. Το 83% της χρηματοδότησης διατίθεται λοιπόν για τον επισητισμό, διότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που αποφασίζουν για το ε, τι χρειάζεται ε, περισσότερο το κάθε κράτος. Στην Πολωνία έχουμε κάνει ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα. Διότι τώρα τα τρόφιμα που διανέμονται είναι βιολογικά, είναι καλύτερης ποιότητας και αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Ενέχεται εδώ και η διάσταση της αξιοπρέπειας. Ο κόσμος έχει έτσι πρόσβαση σε τρόφιμα που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να πληρώσει. Και η έκθεση μας πληροφορεί επίσης ότι έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες να εντοπιστούν οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν ανάγκη από περισσότερη βοήθεια. Υπάρχει μία λίστα κριτηρίων. Αλλά από την άλλη μεριά μας λέτε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, κριτήρια όσον αφορά τα εισοδήματα, να μην κλείνουμε καμιά πόρτα. Τι νομίζετε λοιπόν, θα πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον κατάλογο κριτηρίων ή θα πρέπει το πρόγραμμα να είναι τελείω ανοιχτό, γιατί αυτό εξαρτάται από τον κόσμο, από τι ανάγκε του, από τον τρόπο που δουλεύουν οι μη κυβερνητικέ, οι φιλανθρωπικέ οργανώσει. Δεν νομίζω ότι εδώ μπορούμε να βρούμε μια ενιαία λύση. Θεωρώ λοιπόν ε, πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στους ε, πιο ευάλωτους. Όχι όμως ε, μόνη της. Χρειάζεται συνοδευτικά μέτρα βλέπουμε τα νούμερα και παρατηρούμε ότι ο αριθμός των απόρων στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ψηλός. Και στη χώρα μου έχει σημειωθεί μεν πρόοδος, όμως το πρόβλημα παραμένει. Έχουμε 2% ε, άστεγους στην ε, χώρα μου και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο ταμείο. Βέβαια είμαι σοσιαλδημοκράτης, γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τις, ε, και, να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι κάτι αποκλειστικά τεχνικό. Να δούμε λοιπόν όλες τις προεκτάσεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι η επισητιστική βοήθεια είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε, διότι αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να χτίσουν τα προγράμματα των κρατών μελών, τα οποία αδυνατούν ή να παρέχουν τέτοια βοήθεια ή επικεντρώνονται σε άλλα. Θα χρειαστεί βέβαια να συνεργαστούμε όχι μόνο με το κράτος αλλά και με τους διάφορους μη κυβερνητικού οργανισμούς. και θα πρέπει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση από την επισητιστική βοήθεια ε, στα μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Επίσης, θεωρώ πως ε, θα ήταν ε, καλό να καταπολεμηθούν τα αίτια έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να αγοράζουν μόνοι τους το φαγητό τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. θα μιλήσω σου ειδικά λέει η κυρία Άλσα Εκ μέρους του Ρίνιου ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την έκθεση αυτή. Μερικές φορές με έκπληξη ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο για να έχουν φαγητό στο σπίτι. Και με τη βοήθεια πολλών και τοπικών αρχών και άλλων αρχών θα μπορούσαμε να έχουμε προοδεύσει, να έχουμε βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Ε, μέσω αυτής της προσπάθειας της δουλειάς να καταπολεμήσουμε ε, την ένδυα ε, ίσως θα έπρεπε να σκεπτόμαστε πιο μακροπρόθεσμα διότι το πιο σημαντικό δεν είναι απλώς να μάθουμε πώς να τρώμε ψάρι για παραδείγμα αλλά να μάθουμε πώς να ψαρεύουμε λέει η ομιλήτρια ώστε να μπορούμε να να μπορεί κανείς δηλαδή να θρέψει τον εαυτό του να είναι αυτόνομος εάν θεωρούμε ότι υπάρχει μία άδικη ή άνηση κατανομή πόρων υπάρχουν κάποιες, έχετε εσείς κάποιες συστάσεις αναχώρα πιο συγκεκριμένες. Τι θα μπορούσαν δηλαδή τα κράτη-μέλη να κάνουν ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες τους θα έχουν μια πιο αξιοπρεπή διαβίωση. Δηλαδή νομίζω ότι πιο συγκεκριμένες συστάσεις θα βοηθούσαν και μερικές φορές επίσης θεωρώ ότι καλό είναι να αποφεύγουμε να προσποιούμεθα και να, ότι η κατάσταση είναι πιο ρόδινη. Γιατί υπάρχουν και εντός και εκτός του οίκου αυτού άνθρωποι που ε, όλη τους η προσπάθεια είναι να επικρίνουν και να καταστρέψουν. Ο κύριος ε, Μαγιορίνο, ευχαριστώ την Επιτροπή πρώτα απ' όλα για την ε, ευκαιρία αυτή για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δύο πράγματα ήθελα να αναφέρω απλώς για να είμαι σύντομος. Καταρχάς, ε, όπως μόλις είπε η συνάδελφος, πώς σχετίζονται όλα αυτά με τα υφιστάμενα εθνικά μέσα Δηλαδή πώς συνδυάζεται αυτό το μέσο με τα όσα έχουμε στη διάθεσή μας τα κρατημέλη σε όλα τα επίπεδα. Το δεύτερο και το γνωρίζουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με την περιθωριοποίηση, την κοινωνική, το πιο σημαντικό σήμερα ζητούμενο δεν είναι απλώς να βρούμε καινούριου πόρους, αλλά να μην κατακαιρματίζουμε τους υφιστάμενους πόρους. Γιατί στα διάφορα κράτη-μέλη πάντα έχουμε κάποια μέσα για την καταπολέμηση της ένδυας, είτε εθνικά, κρατικά, είτε κονδύλια δημοτικά, είτε αναλαμβάνοντας ε, πρωτοβουλίες ε, και σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η ελεγχθεί. Επομένως, σήμερα ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, όπου υπάρχει επίγνωση, μεγαλύτερη επίγνωση για την αναγκαιότητα παρέμβασης, η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων παρεμβάσεων. Να μην έχουμε κατακαιρματισμένη προσπάθεια. Και γι' αυτό ήθελα να ακούσω τη σκέψη σας, την άποψή σας επ' αυτού. Και κατά πόσον και υπό την έννοια του κινήτρου θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον για το μέλλον. Δηλαδή να δίνουμε κάποια προώθηση, κάποιο κίνητρο στα μέσα εκείνα τα οποία συντονίζουν καλύτερα τις επιμέρους παρεμβάσει. Ο κύριος Μίλλερ λέει Przewodnicząca. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες και να τους συγχαρώ. Ίσως αυτό που μας λείπει είναι μια λεπτομερής εκτίμηση, ανάλυση των πέντε ετών λειτουργίας του Ταμείου. Γιατί σύμφωνα με την έκθεση η χώρα μας, η χώρα μου η Πολωνία, είναι από τους πιο σημαντικούς δικαιούχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει τα δύο τρίτα των ε, κονδυλίων που δαπανήθηκαν. Ωστόσο, κατά την Πολωνική Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των απόρων στην Πολωνία δεν μειώνεται. Δεν έχει μειωθεί. Και αυτό παρά τους πρόσθετους πόρους που έχουν καταβληθεί από τον εθνικό προϋπολογισμό που έχουν δηλαδή δοθεί σε οικογένειες επί τη βάση των ε, τέκνων οι αυξήσει στα επιδόματα τέκνων δεν έχουν δοκιμαστεί, δεν έχουν ελεγχθεί. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή λαμβάνουν ενισχύσεις άνθρωποι που δεν τις χρειάζονται. Επομένως η ερώτησή μου προς το ελεγκτικό συνέδριο είναι σε ποιο βαθμό οι πόροι του Ταμείου για τους Απόρους πράγματι καταλήγουν στους απόρους, σε εκείνους που έχουν ανάγκη. γιατί από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέρος των χρημάτων αυτών δαπανάται με τρόπο μη αποτελεσματικό. Αν μου επιτρέπετε και εμένα μια ερώτηση, λέει η Πρόεδρος, αναρωτιόμουν για τους διάφορους αριθμούς δικαιούχων που έχετε στα διάφορα κράτη-μέλη. Εγώ είμαι από τη Σλοβακία και έχουμε ένα νομοθετικό ορισμό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ηλική ανάγκη, που, ένδια, απόρους δηλαδή. Και έχουν ανάγκη όχι μόνο χρημάτων, αλλά διαφόρων ενισχύσεων σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι δικαιούχοι και μία από τις προϋποθέσεις είναι η μόνιμη κατοικία. Έχουμε πάρα πολλούς άστεγους ωστόσο. Έχουμε τις ε, κοινότητες των ε, Ρωμά που δεν επίσης εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις. Και σε επίπεδο επιστηστικής βοήθειας υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Ε, υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα και ενδεχομένως πρέπει να πιέσουμε τα κρατημέλη να συμφωνήσουν σε έναν ορισμό κοινό ή τουλάχιστον κοινά κριτήρια, προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα λαμβάνουν βοήθεια επισητιστική ή χρηματική ή άπορη τουλάχιστον σε σχέση με ενωσιακά κονδύλια. Ευχαριστώ. Yes, Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν απαντώντας σχετικά με τη συνεισφορά του ΦΕΑΝΤ στην καταπολέμηση της φτώχειας. Ναι, δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν αρκούν ε, τα στοιχεία της έκθεσης για να οδηγηθούμε σε ε, συμπεράσματα. Αυτό διότι οι μετρήσεις των αποτελεσμάτων ήταν ελλειπείς. Δεν υπήρχαν κάποιοι δείκτες ε, εκείνοι που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Όμως να σας πω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο ταμείο. Από την εμπειρία που έχω με τέτοια προγράμματα είναι ένα οριζόντιο ε, πρόβλημα του ESF, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι δαπάνες ε, γίνονται αλόγιστα όμως υπάρχει δυσκολία ε, στην ε, μέτρηση των αποτελεσμάτων. Ορισμένες φορές είναι απλά τα πράγματα, ξέρεις ότι υπάρχουν αυτά στοιχεία, μπορείς να πας από το α στο β και να ακολουθήσεις τα στοιχεία αυτά. Εδώ όμως η δυσκολία μέτρησης είναι μεγαλύτερη διότι το θέμα είναι πολύπλοκο. Ε, η έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρει ότι από μόνο του το Ταμείο για τους Απόρους δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της φτώχειας. Θα ήταν αστείο αν ε, νομίζαμε ότι 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνδυασμό με άλλα τόσα περίπου εθνικής χρηματοδότησης μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της φτώχειας. Όμως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια προσπάθεια. Φυσικά αναφερθήκατε στο συντονισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ συντονισμός, διότι χωρίς αυτόν όλες οι προσπάθειες από τοπικούς, ε, περιφερειακούς και εθνικούς ε, φορείς ε, θα οδηγήσουν στο πουθενά. Γι' αυτό λοιπόν είναι αδύνατον από μόνο του το ταμείο αυτό να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά σημαντικό, παρότι το ποσό με το οποίο έχει υπηρκοδοτηθεί είναι μικρό, η βοήθεια που παρέχει είναι σημαντική, ιδιαίτερα στον ε, επισητιστικό τομέα, σε αρκετά κρατημέλη. Τώρα, δεν μπορώ να σας πω τον λόγο για τον οποίο κάποια κρατημέλη το χρησιμοποιούν περισσότερο και κάποια λιγότερο. Αυτό εξαρτάται από τα ίδια τα κρατημέλη, διότι ορισμένα επιλέγουν την επισητιστική βοήθεια, ορισμένα επιλέγουν τα μέτρα ε, καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και άλλα πάλι ένα συνδυασμό και των δύο. Όπως ε, σας είπα και πριν, πάνω από το 83% των κονδυλίων του Ταμείου πηγαίνει σε μέτρα επισητιστικής βοήθειας. Ε, τώρα, συμφωνώ απόλυτα για την αξιολόγηση αντικτύπου. Αυτό είναι μια οριζόντια ανάγκη και ε, επικροτώ την πρότασή σας, διότι δίχως αξιολόγηση αντικτύπου, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα φτάσουμε στο στόχο, διότι δεν θα είναι σαφής ο στόχος αυτός. Χρειάζεται λοιπόν να ξέρουμε που βαδίζουμε, να έχουμε ένα μπούσουλα. Να έχουμε γνώση των πραγματικών αναγκών και ε, των ε, πραγματικών ευάλωτων ομάδων. Τώρα, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Συμφωνώ να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε προσπάθειες να παρουσιάζουμε τη συνολική εικόνα της πρόκλησης αυτής. Ε, βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτήν την τάση, για παράδειγμα στην, ε, στο εγγύηση για τους Νέους, να προσπαθεί με λίγα χρήματα να κάνει πολλά, όπως για παράδειγμα με τη, τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Δεν ε, χρειάζονται πολλά χρήματα, αλλά καλή διαχείριση. Τώρα, φυσικά και συμφωνώ με το θέμα της απλοποίησης, αλλά και ε, το θέμα της αηφορίας. Αυτό ισχύει για όλα τα προγράμματα υπό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τώρα, κατανοώ το ότι αρκετοί από εσάς ε, εκπλήσονται με τον αριθμό των ε, απόρων στην Ευρώπη. Και εγώ όταν διάβαζα την έκθεση για να προετοιμαστώ για τη σημερινή παρουσίαση, εξεπλάγει, με σόκαρε το γεγονός ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους δυσκολεύεται είτε να πληρώσει τον νίκη του, είτε τους λογαριασμούς του, είτε ε, σε άλλους ε, τομείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνη. Επίσης, ε, ο ορισμός είναι πράγματι ένα πρόβλημα. Πώς μπορούμε να ορίσουμε την ευάλωτη ομάδα. Πώς μπορούμε να ορίσουμε το τι είναι άπορος, μπορούμε να δούμε κάποιες, κάποιες ομοιότητες, για παράδειγμα με το Ταμείο Εγγύησης για τους Νέους, όπου υπήρχαν κάποια ελάχιστα κριτήρια που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και ίσως αυτό θα έπρεπε να το δούμε για να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ. Βέβαια, το κράτος μέλος είναι εκείνο που θα καθορίσει αυτά τα πράγματα, που θα διατυπώσει τον ορισμό του απόρου. Γιατί φυσικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην σπαταλούμε κονδύλια σε ε, εκείνους που δεν χρειάζεται, τα χρειάζονται. Τώρα, πώς σας είπα, ε, το 83% των ε, κονδυλίων πηγαίνει σε επιστημιστική βοήθεια. Είναι κακό αυτό? Όχι κατά ανάγκη. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου πέντε χρόνια και δεν βρισκόμαστε πια σε αρχικό στάδιο που όλα διαμορφώνονται ακόμα, υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια ερωτηματικά. Συμφωνώ ότι υπάρχουν στοιχεία σχετικά με αυτό που λείπουν από την έκθεση, όμως όταν ξεκινούσαμε τη σύνταξη της έκθεσης ε, μας έλειπαν αυτά τα στοιχεία και για πολλά επιμέρους ε, κομμάτια του προγράμματος έπρεπε να περιμένουμε για να δούμε τα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα την ενσωμάτωση των μεταναστών. Με ρωτήσατε γιατί δεν υπάρχει αναφορά σε αυτό στην έκθεση, διότι η ενσωμάτωση των μεταναστών θέλει χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν ε, ίσως θα ήταν καλή ιδέα να κάνουμε και μία επόμενη έκθεση όπου θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Μετά, έγινε και μία ερώτηση για τη μακροπρόθεσμη εφορία και για το να μάθεις τον άλλο να ψαρεύει από ε, το να του δώσει το φαγητό. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Χρειάζεται ένα συνδυασμός μέτρων για να σημειωθεί πρόοδος. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε από τώρα ε, πως βρήκαμε μια λύση που μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Για παράδειγμα στην ε, Γαλλία και το Βέλγιο ε, τα προγράμματα είναι πιο ευέλικτα, χρησιμοποιούν την επισητιστική βοήθεια με πιο ευέλικτο τρόπο, δεν έχουν τόσο αυστηρά κριτήρια, ενώ σε άλλα κρατημέλη, όπως στη Γερμανία για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τα μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης για την ένταξη των ε, μεταναστών. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον το ότι υπάρχει διαφορετική χρήση των κονδυλίων από χώρα σε χώρα. Τώρα, για τις επόμενες ερωτήσεις, ε, νομίζω πως θα αφήσω ε, χρόνο στο συνάδελφο για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Όπως είπε και η κυρία Ιβάνοβα, εμείς ε, δεν ε, θέλαμε να ελέγξουμε την εφαρμογή του προγράμματο στα κράτη-μέλη. Όχι, εμεί θέλαμε να ε, διεξάγουμε ελέγχους ε, στα ίδια τα προγράμματα. Δεν ε, μπορούσαμε, όπως καταλαβαίνετε, να καλύψουμε όλες τις πτυχέ του θέματος αυτού. Τώρα για την απορρόφηση των κονδυλίων, να πω καταρχάς ότι αυτό είναι ένα οριζόντιο θέμα και ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων ε, κάποιων πληθυσμιακών ομάδων, δεν μπορούμε να έχουμε τόσο καλό έλεγχο όσο θέλουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε ο κάθε δικαιούχος ε, να είναι διαθέσιμος, να μπορεί να απαντήσει σε ερωτηματολόγια και τα λοιπά σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Αυτός ο έλεγχο πρέπει να γίνει σε ανώτερο επίπεδο. Επίση να μην ξεχνάμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν αισθήματα. Μετά, φυσικά είναι και στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους να αποφασίσει ποιο δικαιούται βοήθεια. Ε, είναι και θέμα εθνικής και περιφερειακής ε, πολιτικής, είναι θέμα υποδομών, ε, συνεργασίας με τους συνεργαζόμενους φορείς, με τις διάφορες οργανώσεις που παρέχουν επισητιστική βοήθεια. Μιλάμε για μια μεγάλη αλυσίδα, για διανομή τροφίμων κτλ. Εκεί βοηθά το Ταμείο. Βέβαια, να πούμε ότι το Ταμείο δεν, το κάνει και άλλα πράγματα εκτός από το να παρέχει επισητιστική βοήθεια. Αυτό δεν είναι κριτική είναι γεγονό. Δεν θέλουμε εμείς να ασκήσουμε κριτική στο γεγονό αυτό. Τα προγράμματα και όλα τα συνοδευτικά μέτρα είναι ε, κάτι πρόσθετο στα υπάρχοντα μέσα. Αυτό που μπορούμε με σιγουριά να πούμε είναι ότι αν δεν υπήρχε το ταμείο αυτό, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθετε αυτά τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτή την ε, περίοδο, θα υπήρχαν προβλήματα σε πάρα πολλές οργανώσεις και πολλά κενά. Μπορούμε δηλαδή να καταγράψουμε τις ε, ελλείψεις και τους τομείς όπου χρειάζεται βελτίωση, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, να πω ότι τα κράτη-μέλη ήταν εκείνα που έπρεπε να καθορίσουν το ύψος του, των κονδυλίων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Είχαμε ένα ελάχιστο όριο 3,5 εκατομμύρια ευρώ Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ χαμηλό ποσό, αλλά βοήθησε ε, κατά κάποιον τρόπο τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν το ύψος της ε, βοήθειας. Μετά. Κάτι άλλο. Που ήταν και σύσταση δική μας κιόλας. Κατανοούμε τη σημασία των συνοδευτικών μέτρων, αλλά η κριτική που έχουμε να ασκήσουμε ως ελεκτές είναι ότι δεν είναι συγκρίσιμα, δεν μπορεί να μετρηθεί ο αντίκτυπος των συνοδευτικών αυτών μέτρων. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε διάφορες ευκαιρίες για να γίνει αυτό, ε, διοργανώσε ημερίδες, εκδηλώσεις κτλ. Και τώρα γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα συνοδευτικά μέτρα για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να εντοπιστεί ο κατάλληλος ε, δικαιούχος. Αλλά είναι απλά τα πράγματα. Δίνεις ένα sleeping bag σε έναν άστεγο και αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνεις για να τον βοηθήσεις. Εκεί στοχεύουμε εμείς. Το συνοδευτικό μέτρο όμως είναι ότι μπορείς να τον ενημερώσει, να του πεις ότι μπορεί να πάει σε ε, μια υπηρεσία της πρόνοιας μπορεί να βοηθηθεί και διαφορετικά. Αυτό η κάθε πόλη, η κάθε περιφέρεια πρέπει να το εφαρμόσει μόνη της και αυτό θεωρείται συνοδευτικό μέτρο. Όμως, όταν δίνεις ένα ζεστό πιάτο φαγητό και ένα sleeping bag σε έναν άστεγο είναι μια βοήθεια άμεση και επίσης να μην ε, παραγνωρίζουμε την σημασία των συνεργαζόμενων ε, φορέων και της ε, καλής οργάνωσης. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με συγχωρείτε αν προφέρω καλά το όνομά σας, κύριε Πιετραντώνιο. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι και εγώ τις εκτιμήσεις σας. Μ' αρέσουν πολύ οι εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου, διότι περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία, πληροφορίες και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη βοήθεια που παρέχουμε. Το σημαντικό με το ηλεκτρονικό συνέδριο είναι ότι δίνει αρκετές ε, απαντήσεις ε, και πληροφορίες. Κάνει, αν θέλετε, συμπληρωματικό εργοστάσιο σε αυτό που κάνουμε εμείς. Τώρα, πρόκειψαν κάποια θέματα, κυρίως επιλεξιμότητας. Ποιος είναι επιλέξιμος ε, στοχεύουμε στις κατάλληλες ομάδες, επιλέγουμε τους ε, σωστούς δικαιούχους. Αυτό πρέπει να το δούμε και από το, υπό το εθνικό πλαίσιο. Η επιλεξιμότητα βέβαια είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, ιδιαίτερα ε, αν αναλογιστεί κανείς την επικουρικότητα. Βέβαια πρέπει να σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όταν... Ε, επιλέγουμε τις, ε, τους δικαιούχους. Βέβαια, η νέα πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ συμπεριλαμβάνει και κάποια στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν με τη σειρά του στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όμως επαναλαμβάνω ότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που καθορίζουν ε, την επιλεξιμότητα. Τώρα, χρειάζεται τα μέτρα να είναι και συμπληρωματικά. Και να σας ενημερώσω ότι ο κανονισμός ε, για το Ταμείο έχει απλουστευτεί κατά πολύ σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό την επιμερισμένη διαχείριση. Για τις ε, επιμέρους δυνατότητες και στόχους του ΦΕΑ. Τους στόχους 10 και 11 έχουν γίνει σημαντικές απλουστεύσεις σε ό,τι αφορά τους δείκτες, την ε, υποβολή εκθέσεων, τον ε, επιμερισμό του ε, φόρτου και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς. Όπως είπε και ο αγαπητός κ. Λούπλο, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρέπει να ε, προσέχουμε και τις ε, μεμονωμένες ε, περιπτώσεις. Πρέπει να κοιτάμε τον άνθρωπο. Η εκτίμηση κοινωνικού αντικτύπου είναι κάτι που χρειάζεται επίσης. Έχει γίνει εξάλλου στο παρελθόν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό τα προγράμματα να ξεκινούν από τη βάση όταν τα κράτη-μέλη καταρτίζουν διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα, πρέπει να παρέχεται και μια δυνατότητα παρέμβασης, η οποία θα διέπεται από ένα σκεπτικό φυσικά. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ προσεκτικοί στην εφαρμογή των επιμέρους στόχων. 10 και 11. Να ολοκληρώσω ότι και να πω ότι η ψηφοφορία της, προηγου... της ε, προηγούμενης επιτροπής για το ESF ε, Plus μας ε, ικανοποίησε πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχίσει και με αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας. Καλή τύχη με τις επόμενες εκθέσεις. Όπως σας είπα και πριν, ε, εκτιμώ πάρα πολύ το έργο σας. Ε, μ' αρέσει να βλέπω συγκεκριμένα στοιχεία, δεδομένα και αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα βέβαια είναι ένας προβληματικός ε, τομέας, διότι πάντα κοιτάμε τα νούμερα. Και πιστεύω πως δεν κάνουμε σωστά, διότι μόνο με νούμερα δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ σταματάει η συνεδρίαση. Καλή όρεξη σε όλους και θα σας δω το απόγευμα στην ακρόαση της κυρίας Ντάλη.